Okay, friends. Um... Ε, αγαπητοί φίλοι, ξεκινούμε και πάλι οικονομικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2018 Σε στάσει αναχώρα. Καλώς ορίζουμε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Οικονομικό Διάλογο Αρμόδιο και την κυρία Τίσεν Αρμόδια για τα θέματα των ε, κοινωνικών ζητημάτων, ε, ε, δικαιωμάτων των εργαζομένων, κινητικότητα των εργαζομένων. Σε ευχαριστούμε που είναι εδώ. Έχουμε την ανταλλαγή απόψεων για τις συστάσεις αναχώρα. Δυστυχώς ο Επίτροπος Μασκοβισσή αρμόδιος για τα οικονομικά και δημοσιονομικά, φορολογικά και τελωνιακά ζητήματα, δεν μπόρεσε να έρθει, ακύρωσε χθε το βράδυ την ε, συμμετοχή του στη σημερινή συζήτηση λόγω διάφορων εξελίξεων συναφών με το Συμβούλιο, όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που λαμβάνει η χώρα σήμερα και αύριο. Η Επιτροπή θα μας παρουσιάσει λοιπόν τις εκθέσεις αναχώρα και την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με τα, προγράμματα, εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και ε, σταθεροποίησης που προγραμματίζεται να υιοθετήσει το Συμβούλιο στις 13 Ιουλίου και τα οποία στη συνέχεια καλούνται τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν εφαρμόζοντας τις συστάσεις αυτές, στις δημοσιονομικές, τους εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές το 2018-2019. Με βάση λοιπόν τα Ιωθώτα και το χρόνο που δίνουμε για τη συζήτηση και τις ερωτήσεις. Το πρόγραμμα είναι ως εξής. Θα γίνουν εισαγωγικές παρατηρήσεις 15 λεπτών εκάστου συνολικά, μάλλον 15 λεπτών συνολικά, αλλά μια και δεν είναι εδώ ο κ. Μοσκοβίση, μπορούμε να το επεκτείνουμε λίγο αυτό. Μετά θα ακούσουμε τις ερωτήσεις και παρατηρήσεις των συναδέλφων τη Επιτροπής μας. Θα δώσουμε μετά το περιθώριο στην κυρία Τίσεν και κάποιους βουλευτές. Που σε μισή ώρα περίπου θα χρειαστεί να αποχωρήσουν για την τελετή υπογραφής της οδηγίας για την απόσπαση εργαζομένων, οπωσδήποτε πολύ σημαντικό στόχος και έτσι δεχόμαστε την διακοπή αυτή. Στα Σταματώ εδώ και δίνω το λόγο στον κύριο Ντομπρόφσκης. Έχετε το λόγο. Και σε, περιμένουμε να ακούσουμε με πολύ ενδιαφέρον τα λόγια σας. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να έρθω σήμερα εδώ μα με την Επιτροπή για να παρουσιάσω τι συστάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι ε, οικονομικέ πολιτικέ των επόμενων 12-18 μήνων, όπω τι υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται να τι υιοθετήσει ε, το Συμβούλιο αυτή την εβδομάδα για να τις επικυρώσει τον Ιούλιο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με προτεραιότητες, ε, δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις και υπεύθυνε δημοσιονομικές πολιτικές. Έχουμε τα, τις προτάσεις αναχώρα και τα επίπεδα ε, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη περιγράφονται σε αυτές και βέβαια υπάρχουν και ειδικέ συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ Στηριζόμαστε επίσης στον Ευρωπαϊκό κοινώνα, Επιλώνα Κοινωνικών ε, Δικαιωμάτων για τον εξυγχρονισμό των ε, συστημάτων ε, απασχόληση και κοινωνική προστασία, που θα σα εξηγήσει η Μαριάννη. Ιδιαίτερη έμφαση έχουμε δώσει στον κοινωνικό διάλογο και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταιρών ε, στην διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων. Έχουμε ενισχύσει το διάλογο με το, τις εθνικές αρχές, ε, τα κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους, όλους του εμπλεκόμενου ε, φορεί, ιδιαίτερα δίνουμε έμφαση στον δημοκρατικό διάλογο και οπωσδήποτε προσωπικός τιμώ ιδιαίτερα την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Κάθε επίπεδο εθνικό κτλ. είναι ένα επίπεδο πολύ σημαντικό για τον διάλογο και για όλους μας εδώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συστάσεις μας καταφθάνουν σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό και οικονομικό κλίμα με ταχύτερη από όλη τη δεκαετία ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας που αναμένεται να συνεχιστεί έστω και με λιγότερο ταχύς ρυθμούς. Ανάπτυξη, επενδύσεις, δημοσιονομικά όλα έχουν θετικές ε, τάσεις. Οι μακροοικονομικές ισορροπίες έχουν προχωρήσει, ωστόσο το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος αλλά και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διατηρούν υψηλά ποσοστά σε άκρητα σε αρκετά κράτη-μέλη, προστατευτισμός ε, ελοχεύει στην παγκόσμια αγορά και βλέπουμε επίσης μία άνηση αντίδραση ανατομής και χώρες ως προς τις δικές μας συστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν, μια και είναι ευνοϊκή η συγκυρία, πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε για να ευνοήσουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση. Διαρθρωτικές αλλαγές για να αντιμετωπιστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες για να έχουμε ένα περιθώριο στην προσεχή αρνητική συγκυρία, βελτίωση του περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις ε, ε, και ιδιαίτερα για το άνοιγμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα σε πολλές ε, χώρες, βελτίωση της διακυβέρνησης, αντιμετώπιση της διαφθοράς, συνεχείς προσπάθειες για τον εξυγχρονισμό της αγοράς εργασίας και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, βιωσιμότητα των σταξιδοτικών ε, και συστημάτων ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για ορισμένα κράτη, που όμως θα είναι ούτως ή άλλως πρόκληση για όλα τα κράτη-μέλη. Προτάσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης και κυρίως των δεξιοτήτων μέσα από την ε, μαθησιακή διαδικασία και την κατάρτιση και τη διαβίου μάθηση, αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων είναι η προτάση μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα κύριο μέλημα την εξασφάλιση μιας στεναρής και ανθεκτικής οικονομίας για κάθε χώρα, γιατί ό,τι μπορεί να συμβεί στη μία χώρα επηρεάζει και τις άλλες. Πρέπει να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, ανθεκτικές, αλλά και ανοιχτές σε όλους οι οικονομίες μας και γι' αυτό τα προγράμματα διαρθρωτικών, ε, διαρθρωτικής υποστήριξης για την περίοδο μέχρι το 2020 ενισχύονται και προσαρμόζονται αντιστοίχω και για την περίοδο μετά το 2020 και ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσετε και εσείς να μας υποστηρίζετε. Ε, το, το σύμφωνο ε, ανάπτυξη σταθερότητας που υποστήριξε την προηγούμενη εβδομάδα το, Ευρω... το Συμβούλιο προτείνει τα μέτρα αυτά έχουμε ε, διακοπή του, προγράμματος υπερβολικού ελλείμματος για τη Γαλλία, καθώς μείωσε το έλλειμμα της η Γαλλία κάτω από το 6% και έτσι μένει μόνο η Ισπανία στην ε, διορθωτική ε, προσέγγιση από τις 23 χώρες που είχαμε το 2011. Έχει κάνει τις προτάσεις ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσαρμόζεται με το σχέδιο, το διορθωτικό σχέδιο προϋπολογισμού η, Ευρωπαϊκή, η Ισπανική κυβέρνηση. Αντίστοιχα και ο, η Γερμανική ε, κυβέρνηση έχει κάνει προτάσεις σύμφωνες με το σύμφωνο. Συμμόρφωση έχουμε και με την Ιταλία και με το Βέλγιο προς τα κριτήρια του χρέους Υπήρξε η πρόταση για άνοιγμα διαδικασίας ε, υπερβολικού χρέους, αλλά διακόπτεται αυτή τη στιγμή. Σημαντικές είναι οι αποφάσεις που αφορούν την ε, Ρουμανία και την Ουγγαρία. Έχουμε επίσης έκθεση προσαρμογής διετή με βάση τα κριτήρια σύγκλησης και την, ανταγων... και την συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας ως προς το ευρωπαϊκό δίκαιο για το ευρώ. Από τις 7 χώρες που εξετάσαμε, καμία δεν πληρεί όλους τους όρους του ευρώ. Βουλγαρία, Κροατία, Σουηδία, μόνο σε ονομαστικούς όρους, πλην της ε, σταθερότητας των ισοτιμιών, που θα πάει στον ε, μηχανισμό σταθερότητας επίσης. Η δε Κροατία είναι απολύτως ε, συμμορφωμένη στο θέματα της Ευρωζώνης με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έτσι λοιπόν, η συνεργασία σε όρους οικονομικούς και νομισματικούς σε μια νομισματική ένωση, η οικονομική ένωση δεν είναι θέμα επιλογής, είναι αναγκαιότητα, είναι αδύρυτη ανάγκη και ως εκ τούτου αυτή η ε, οικονομική ένωση μπορεί να προχωρήσει μόνο όταν όλες οι χώρες συμμορφωθούν και συνεργαστούν στο ίδιο επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο κατευθείαν στην κυρία Τάισεν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, όπως είπε ο Βάλτης, η οικονομία αναπτύσσεται με τους γρηγορότερους ρυθμούς που έχουμε δει την τελευταία δεκαετία και αυτό σημαίνει ότι τώρα έχουμε την ευκαιρία να κοιτάξουμε πιο μπροστά και να δημιουργήσουμε μια βάση για βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Επίσης είναι η κατάλληλη στιγμή να έχουμε ε, δημοσιονομικές εγγύσεις για να μετριάσουν ε, τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις ε, μελλοντικών κλειδονισμών. Σχεδόν 238 εκατομμύρια εκατομμύρια Ευρωπαίων είχαν θέσει απασχόλησης και 7,1 είναι η συνολική είναι η ανεργία, πλησιάζει δηλαδή τα επίπεδα πριν την κρίση και οι μεταρρυθμίσει που έχουν εισάγει τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια ε, έχουν αποφέρει καρπούς. Η οικονομική ανάπτυξη όμως δεν ωφελεί όλους τους πολίτες. Η ανεργία παραμένει υψηλή σε κάποιες χώρες, στην Ελλάδα 21%, 17% στην Ισπανία. Είναι υψηλή σε κάποιες περιφέρειες και είναι και υψηλή σε κάποιες ομάδες, ιδιαίτερα τους νέους σε κάποια κράτη-μέλη. Οι ανισότητες ε, είναι ακόμα κάπως αυξημένες σε σχέση με πριν την κρίση και δεν έχουμε σταθερότητα τα τελευταία χρόνια. Είδαμε αύξηση σε κάποια κράτη-μέλη από το 2010 και μετά παρόμοια τάση βρίσκουμε όσον αφορά τους ανθρώπους που κινδυνεύουν από φτώχεια. 23% αυτή τη στιγμή στην Ένωση, η αύξηση έχει σταματήσει, αλλά ακόμα απέχουμε από τους στόχους μας ε, στο πρόγραμμα Ευρώπη 2020 και κάποια κράτη-μέλη έχουν δει σημαντικές αυξήσεις από το 2010 και μετά. Για τους λόγους αυτούς είναι σημαντικό να συνεχιστούν οι προσπάθειες μας για μεταρρύθμιση και να συμβάλλουν όχι μόνο στην οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την κοινωνική δικαιοσύνη, την ε, σύγκληση και την ε, ε, κοινωνική κινητικότητα προς τα επάνω. Ο κοινωνικός πυλώνας δικαιωμάτων, καθώς και ο πίνακας αποτελεσμάτων, μας είναι εργαλεία για μας ε, για να τα πετύχουμε αυτά. Και έχουμε συστάσεις αναχώρα φέτος ε, με επίκεντρο ε, την απασχόληση, την εκπαίδευση και κοινωνικά θέματα. Θέλουμε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη να φροντίσουμε η οικονομική ανάπτυξη να συνοδεύεται από κοινωνική ανάπτυξη. Ο γρήγορος ρυθμός ε, της τεχνολογικής προόδου περισσότερο από ποτέ απαιτεί προσπάθειες ε, για την ε, αναβάθμιση των δεξιοτήτων των Ευρωπαίων εργαζομένων και να και η ίση πρόσβαση σε εκπαίδευση ποιότητας θα έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες και για τα άτομα που αφορά, αλλά και για την κοινωνική συνοχή και ευημερία των κοινωνιών μας. Η εκπαίδευση των εργαζομένων στην αγορά εργασίας ε, αποτελεί το κλειδί Υπάρχουν διάφορες ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι μετανάστες, ε, τα άτομα με ειδικέ ανάγκες, οι ε, Ρώμα συναντούν υπερβολικά πολλά εμπόδια. Η δυνατότητα να συμμετέχουν στην κοινωνία θα πρέπει ε, να δίδεται εξίσου σε άντρες και γυναίκες. Το να ξεκινήσει κανείς η οικογένεια δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος της κοινωνικής και εργασιακής ζωής. Γι' αυτό οι κοινωνικές υπηρεσίες είναι απαραίτητες. Θέλουμε επίσης να δούμε περισσότερες γυναίκες να εργάζονται. Θα πρέπει να σπάσουμε επίσης ε, το ε, γυάλινο ταβάνι που υπάρχει, το, αυτό που εμποδίζει τις ε, γυναίκες να έχουν υψηλές θέσεις. Υπάρχει σημαντική ανισότητα στο εισόδημα και Πρέπει κάποια κράτη-μέλη να προσέξουν ιδιαίτερα την ε, ανακατανομή ε, των χρημάτων για να αποφύγουμε την ε, φτώχεια. Θα πρέπει δηλαδή να έχουμε σωστή κοινωνική ασφάλιση. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ποιότητας στον τομέα της υγείας. Κυρίες και κύριοι, κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Ευρωβουλευτές για την ε, συμβολή τους ε, στην ε, υιοθέτηση της νομικής πράξης για τις κατευθυντήρες γραμμές για την απασχόληση. Επίσης, με τον συμβιβασμό τονίζουμε περισσότερο τις ίσες ευκαιρίες στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τις δίκαιες συνθήκες εργασίας και την κοινωνική προστασία και ένταξη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Thank Εμείς ευχαριστούμε. Τώρα, υπάρχει δυνατότητα για ερωτήσεις. 1,5 λεπτό η κάθε ερώτηση προς τους ε, επιτρόπους. Και θα αρχίσουμε με το ΕΛΚ, Επιτροπή Απασχόλησης. Ο κύριος Κρίστοφ Χέτμαν. Είσαστε εδώ? Ναι. Ναι, ναι, εδώ είμαι. Α, ναι. Ωραία. Καλώς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θέλω να μιλήσω πολωνικά παρακαλώ, οπότε χρησιμοποιήστε τα ακουστικά σας για να με καταλάβετε. Αγαπητοί ε, Αντιπρόεδρε, αγαπητοί ε, κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βλέπουμε ότι έχει ανακτήσει μια κάποια ταχύτητα η ευρωπαϊκή οικονομία σε όρους δημοσιονομικούς, απασχόληση επενδύσεων που παρουσιάζουν θετική εικόνα. Ωστόσο, θέλω να σημειώσω ότι και η μείωση της ε, ανεργίας δεν αρκεί. Δεν μπορούμε να ε, επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας, ιδιαίτερα για την ανεργία των νέων. Γιατί ο κατακαιρματισμός της αγοράς ε, εργασίας, φτώχεια των εργαζομένων ή εργαζομένων που παραμένουν φτωχοί, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης ε, και κοινωνικής πρόνοιας ε, πρέπει να ε, εξασφαλίσουν μια αγορά πλήρη εργασίας, μια αγορά ολοκληρωμένη, η οποία θα εξασφαλίζει καλές συνθήκες απασχόλησης για όλους. Με κατάλληλη κοινωνική προστασία ακόμα και αν πρόκειται για μη συμβατικούς τύπους εργασίας. Πρέπει να τονίσω επίσης ότι αλλάζει αλλάζουν οι μορφές της εργασίας λόγω της ψηφιακής τεχνολογίας και άρα πρέπει και αυτό να το καλύψουμε. Πρέπει επίσης να ευνοηθεί η κινητικότητα των εργαζομένων, η δυνατότητα εισόδου και εξόδου από την αγορά εργασίας να διευκολυνθεί, να εξασφαλίζεται καλύτερο συνδυασμός επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, να υπάρχουν οι συνθήκες ώστε οι γονείς να μπορούν να εργάζονται ξέροντας ότι τα παιδιά τους την χάνουν της κατάλληλης μέρημνας σε βρεφονιμπιακούς σταθμούς επί παραδείγματι. Ε, και εδώ αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι δεν έχουμε πάντα την ε, ε, αρμονία που χρειάζεται στην αγορά εργασίας. Δηλαδή δεν έχουν καλυφθεί όλα τα ζητήματα ε, παρά κάποιες πρόοδους που σημειώνονται που χρειάζεται ο εργαζόμενος για να μπορεί να ε, είναι ικανοποιημένος μέσα στην αγορά εργασίας. Ερωτώ λοιπόν οι συστάσεις αυτές με ποιο στόχο προχωρούν, με ποιο σχέδιο εσείς θα ενθαρρύνετε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην τήρηση των ε, ε, συστάσεων. Και βεβαίω οι διερμηνεί υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά ότι τα κείμενα είναι γραπτά, διαβάζονται με ταχύτητα του ρυθμού και είναι πολύ δύσκολο να τα ακολουθήσουμε. Παρακαλώ, εσείς τώρα έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε. Ε, μία μου ερώτηση θα ήταν για τον Επίτροπο Μοσκοβισή, αλλά δεν είναι εδώ, οπότε θα το ρωτήσω εσάς, ε, κύριε Τεμπρόφσκι. Η πρώτη μου έχει να κάνει με τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Στις 18 ε, Ιουνίου έγιναν κάποιες προτάσεις για το 2019. Θα συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την περιγραφή των περιοριστικών fiscal stands που περιλαμβάνει η έκθεση για, με την πρόταση για το 2019. Και τι αλλαγές προτείνονται πιο συγκεκριμένα ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη επέκταση και όχι περιορισμός. Στην πράξη επίσης πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Το δεύτερο για το φορολογικό ήταν, όπως σας είπα για τον Επίτροπο Μοσκοβισή, υπάρχει ένα νέο στοιχείο στο ευρωπαϊκό εξάμεινο και είναι η επιθετική ε, φορολογική πολιτική. Εμείς θέλουμε να αντιμετωπίσουμε συντονισμένα τις ε, κακές πρακτικές. Πώς θα γίνει για να, να βοηθήσουμε σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έπρεπε να έχει ένα συντονιστικό ρόλο και κάτι ακόμα. Η ομάδα του κώδικα δεοντολογίας για τις χώρες μέλη αυτό το ρόλο δεν θα έπρεπε να είχαν το συντονιστικό. Οπότε ρωτάω τους επιτρόπους. Ναι, ή όχι. Τι λέτε για αυτό τον κώδικα θετολογίας. Πιστεύετε ότι θα κάνει αυτό το συντονιστικό έργο ή δεν μπορεί, οπότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βοηθήσει κάπως αλλιώς να γίνεται αυτός ο συντονισμός. Ευχαριστώ. Παρακαλώ ο κύριος Στοβροφσκής να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Για τις πρώτες ερωτήσεις μιλήσατε για πολλά και διάφορα θέματα στο κοινωνικό τομέα και σε αυτά θα απαντήσει σίγουρα η Μαριάννα. Αλλά εγώ θα μιλήσω περισσότερο για την υλοποίηση των ε, αναχώρα συστάσεων. Πράγματι, όπως είπα και πριν, υπάρχει πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση των συστάσεων αυτών, αλλά είναι άνηση μεταξύ των χωρών μελών και μεταξύ διαφορετικών τομέων πολιτικής. Βλέπουμε σε μερικές περιπτώσεις να υπάρχει περιορισμένη υλοποίηση, αλλού μεγαλύτερη. Έχουμε βέβαια μια κλίμακα, μιλάμε για καθόλου πρόοδο, λίγη πρόοδο, αρκετή πρόοδο, ουσιαστική πρόοδο κλπ. Βλέπουμε πράγματι ότι μπορούν να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Οπότε λέτε, με ποιους τρόπους μπορούμε να διασφαλίσουμε την υλοποίηση των συστάσεων. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να υπάρξει μεγαλύτερος ενστερνισμός των συστάσεων αυτών σε εθνικό επίπεδο. Εξού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτενώς έχει συζητήσει με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με τις κυβερνήσεις, με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ε, εμπλεκόμενους στις χώρες μέλη. Συζητάμε μαζί τους και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τις συστάσεις αναχώρα, απαντάμε στις ερωτήσεις τους έτσι ώστε να ε, μπορέσουν να ταυτιστούν περισσότερο και να καταλάβουν καλύτερα τις προκλήσεις και έτσι να βοηθήσουν και με λύσεις. Δεύτερον, κάτι που προτείνουμε τώρα για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλαδή μετά από το 2020, είναι να διασφαλίσουμε και μια πιο άμεση σύνδεση ανάμεσα στις συστάσεις αναχώρα και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Με την ευρεία έννοια, δηλαδή διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις επίσης και νέες μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε με 25 δισεκατομμύρια ευρώ τα περισσότερα χρήματα θα πάνε στο εργαλείο επιδόσεων μεταρρυθμίσεων. Προκειμένου δηλαδή να δοθούν οικονομικά κίνητρα στις χώρες ε, μέλη για να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις αυτές. Και το πρώτο σημείο αναφοράς βέβαια είναι το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και οι συστάσεις αναχώρα. Τώρα έρχομαι στην Δεύτερη ερώτηση για τον προπολογισμό για την Ευρωζώνη. Είχαμε ανταλλαγή απόψεων στο Fiscal Board, όντως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την σύσταση αυτή να υπάρξουν πιο περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα. Ε, συζητήσαμε λοιπόν για την Ευρωζώνη, αλλά βλέπουμε ότι η οικονομία εξακολουθεί να επεκτείνεται. Είμαστε στο έκτο έτος μεγένθησης, οπότε μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε καλούς οικονομικούς καιρούς και συνεπώς είναι πολύ καλό να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα μέτωπο εγγύσεων προστασίας ώστε να έχουμε περισσότερα περιθώρια αν κάποια στιγμή τα πράγματα πάνε χειρότερα. Εμείς στηρίζουμε την λογική αυτή του Συμβουλίου να περάσει σε κάπως πιο περιοριστικά fiscal stance. Πάντως οι αποφάσεις σε αυτό το τομέα δεν έχουν ληφθεί. Έτσι κι αλλιώς θα αποτελέσουν ε, μέρος του κύκλου του φθινοπόρου για το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Τώρα για τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό που με ρωτήσατε και αυτό είναι μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πράγματι, θέματα που έχουν να κάνουν ε, με αυτό τα βάζουμε στις εκθέσεις μας αναχώρα και το έχουμε κάνει για 7 χώρες μέλους. Γιατί το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ε, τι είναι, πρόκειται και για το συντονισμό της δημοσιονομικής και της μακροοικονομικής πολιτικής και η φορολογία πάντα ήταν μέρος ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Αν δείτε τις συστάσεις αναχώρα θα δείτε ότι υπάρχουν τέτοιες συστάσεις για πολλές χώρες φορολογικού τύπου. Όσον αφορά αυτόν τον επιθετικό λοιπόν φορολογικό σχεδιασμό και αυτό αποτελεί μέρος της οικονομικής και κοινωνικής μας ατζέντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η φορολόγηση σε εθνικό επίπεδο ε, μπορεί να πλήττει τον ανταγωνισμό και έχει και επιπτώσεις και εκτός συνόρων μιας χώρας, ακόμα και αν είναι θέμα εθνικό. Οπότε ασχολούμαστε και με αυτό το θέμα, φορολογικό σχεδιασμός είναι και αυτός μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Μαρία Αρένα. Ευχαριστώ πολύ. Ω σοσιαλιστές και δημοκράτες χαιρόμαστε βέβαια που βλέπουμε στα πλαίσια των αναχώρασης τάσεων να συμπεριλαμβάνεται και μια πιο κοινωνική διάσταση και θέματα τα οποία υπάρχουν στον κοινωνικό πυλώνα. Όμως διαπιστώνουμε ότι το εξάμεινο κυρίως επικεντρώνεται στο οικονομικό σκέλος και όχι αρκετά στο κοινωνικό. Σήμερα βρισκόμαστε πάντα σε αυτό το πλαίσιο. Μιλάμε για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως μπορεί να είναι αντιπαραγωγικές όταν μιλάμε για κοινωνικούς στόχους. Τι εννοώ? Ευελιξία στο χώρο της εργασίας μπορεί να καταλήξουμε σε μια διαφορετική μεταρρύθμιση όσον αφορά την ευελιξία στην εργασία και να βρούμε πολλά αρνητικά για εργαζόμενους που είναι πιο ευάλωτοι. Συνεπώς, η πρώτη μου ερώτηση είναι πώς εκτιμάτε τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα, δηλαδή μία ε, διαφορετική μεταρρύθμιση θα πρέπει να τη δούμε, να δούμε και τι κοινωνικές επιπτώσεις έχει. Γιατί προς το παρόν αυτό που κάνουμε είναι κοιτάμε πόσα θα εξοικονομήσουμε από αυτήν και όχι τι κοινωνικές επιπτώσεις μπορεί να έχει. Γιατί μπορεί μειώνοντας τις δαπάνες για την υγεία να περιορίζουμε κάπως τις δαπάνες, αλλά στο κοινωνικό τι επιπτώσεις έχει αυτό. Οπότε πώς βλέπετε εσείς τις διαφορετικές αυτές μεταρρυθμίσεις υπό τοπτικό πρίσμα ε, της κοινωνικής παραμέτρου. Έπειτα η σταθερότητα είναι κάτι που πλήρωσαν οι εργαζόμενοι και οι πιο ευάλωτοι στις κοινωνίες μας. Και λιγότερο πλήρωσαν γι' αυτό οι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί. Μπορείτε εσείς να μας πείτε ποιο είναι το κόστος της ε, σταθερότητας αυτής και ποιος τελικά την πλήρωσε γιατί σήμερα υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι τη μέση εργατική τάξη, η οποία ξέρει ότι αυτή πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά τι μεταρρυθμίσεις και επιπλέον βλέπει ότι οι υπηρεσίε που είναι στη διάθεσή της σήμερα στην Ευρώπη είναι χαμηλότερης ποιότητας. Αν θέλουμε λοιπόν να λύσουμε το πρόβλημα αυτή τη δυσαρέσκειας στην Ευρώπη, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ακριβώ αυτό δώσατε κάποια αποτελέσματα για την ανάπτυξη, που είναι θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη μεγένθηση. Αλλά να δούμε πιο συγκεκριμένα, και έχουμε συστάσεις αναχώρα, αλλά εγώ θα ήθελα να έχουμε και μία προσέγγιση περιφερειακή. Υπάρχει τέτοια περιφερειακή για το αν αυξήθηκαν οι ανισότητες, αν υπάρχει ε, μικρότερη σταθερότητα τώρα στην απασχόληση, κοινωνική δικαιοσύνη κτλ. Νομίζω ότι θα έπρεπε και εδώ να έχουμε απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσέγγιση να μην είναι συνολική, όλα πάνε καλύτερα, ορίστε δείκτες είναι θετικοί όσον αφορά τη μεγέθυνση, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα δυσκολίες και αυτές τις δυσκολίες πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ακόμα. Πρόεδρο, σε ευχαριστώ. Ωραία, θα αρχίσουμε αυτή τη φορά με την κυρία Τάισεν να απαντήσετε όλες τις ερωτήσεις που ακούστηκαν μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ για τις Ερωτήσει σας. Θα απαντήσω στα Ολλανδικά, μια που έχουμε εξαιρετική διερμηνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και την αιτήσια αυτή η άσκηση, το χείρημα, πρέπει να σας πω ότι ακόμα και από τα συνδικάτα ξέρουμε ότι το εξάμεινο του 2018 είναι το πιο κοινωνικό εξάμεινο που είχαμε ποτέ. Οπότε νομίζω ότι τη βλέπουμε την εξέλιξη από τότε που ξεκινήσαμε τη θητεία μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το 2014 δηλαδή μέχρι σήμερα, ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ότι όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο κοινωνικό είναι αυτό το εξάμεινο και όλο και πιο ισορροπημένο. Βέβαια, διαρθρωτικά το βλέπουμε, ναι, μαζί αναπτύξαμε τον κοινωνικό πυλώνα, που χωρίζεται σε τρία κομμάτια και προσπαθούμε έτσι να τροφοδοτήσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο και με κοινωνική διάσταση. Κατευθύνσεις γραμμέ για την απασχόληση, για παράδειγμα, που αναφέρεται στις, συστάσεις, σε εκθέσεις μάλλον αναχώρα. Και όσον αφορά τις συστάσεις, και αυτές εμπνέονται από τα αποτελέσματα του κοινωνικού βαθμολογίου που προβλέπει ο κοινωνικό πυλώνα. Άρα, όλο και περισσότερο λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική διάσταση. Τώρα, για τι μεταρρυθμίσει στι χώρε μέλη, που πρέπει να γίνουν περισσότερα, εννοείται έτσι είναι. Όσον αφορά τα δημόσια οικονομικά, υπάρχει βελτίωση, αν συγκρίνουμε το 2014 με το 2017 με το 2018. Υπάρχει τεράστια πρόοδος, αλλά η σταθερότητα των δημοσίων οικονομικών είναι κάτι αναγκαίο. Χρειάζεται, είναι απαραίτητο. Αλλιώς είμαστε σε κίνδυνο για το μέλλον. Εξού λοιπόν και ε, δουλεύουμε περισσότερο για την ε, Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Από εκεί και πέρα χρειάζεται ευθύνη των χωρών μελών. Πρέπει να δούμε ποια είναι η ποιότητα των ε, δημοσίων δαπανών. Και όσον αφορά την κοινωνική διάσταση, βλέπουμε τι πάει καλά, τι πάει λιγότερο καλά. Και βλέπουμε ότι πράγματα όσον αφορά τι ανισότητε, σε πολλέ χώρε εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά την κοινωνική ένταξη και στην αγορά εργασίας και στην εκπαίδευση και εκεί υπάρχουν μερικές φορές σοβαρά προβλήματα. Τα ξέρουμε, τα εντοπίζουμε, ξέρουμε σε ποιες χώρες υπάρχουν προβλήματα περισσότερο από ό,τι αλλού. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει βελτίωση. Εννοείται. Το είπαμε, να έχουμε διάλογο με τις χώρες μέλη, με τους κοινωνικούς εταίρους, με την κοινωνία των πολιτών. Είναι μια διαδικασία διαλόγου που υπάρχει και γίνεται με τις χώρες μέλη. Επίσης, πιέζουμε τις χώρες μέλη να κάνουν περισσότερα, να χρησιμοποιήσουν τα διορθωτικά ταμεία, την τεχνική αρρωγή που προσφέρουμε. Και έτσι προσπαθούμε να πιέσουμε υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Δεν δουλεύουμε δηλαδή μόνο από μόνοι μας και να ξέρετε ότι δουλεύουμε και με τον ΩΣΑ. Και πολλές χώρες ε, στα πλαίσια του ΩΣΑ βοηθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από στρατηγικά σχέδια ώστε να υπάρξει καλύτερο επίπεδο μεταρρυθμίσεων. Επίσης έχουμε και τους ε, στόχους για τα επαγγελματικά προσόντα. Για όλα αυτά προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις χώρες για να πετύχουν μία σταθερή ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Προσπαθούμε να υπάρχει περισσότερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας και των πιο ευάλωτων ατόμων, είτε πρόκειται για ε, άτομα με αναπηρίες, είτε πρόκειται για μετανάστες. Μας ενδιαφέρει. Καταλαβαίνουμε ότι κάποιες κατηγορίες έχουν λιγότερες πιθανότητες ένταξης στην αγορά εργασίας και γι' αυτό προσπαθούμε και βοηθούμε τις χώρες μέλη. Το είπαμε και στην αρχή. Από τις ε, αναχώρας συστάσεις οι περισσότερες υλοποιούνται, γίνονται μεταρρυθμίσεις με επιτυχία, περισσότερο ή λιγότερο προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό ισχύει για τις μισές περίπου, αν δούμε μεσοπρόθεσμα. Μακροπρόθεσμα υπάρχει μεγαλύτερη ακόμα επιτυχία. Αλλά βέβαια είναι πράγματα όπως ε, η εκπαίδευση, υγεία που αλλάζουν πιο αργά. Εμείς στηρίζουμε τις χώρες μέλη με τεχνητή αρρωγή, με τα διαφορετικά ταμεία και ελπίζουμε κάθε χρόνο να έχουμε βελτίωση. Υπάρχουν δυσκολίες ακόμα, πρέπει να το παραδεχτούμε, αλλά πρέπει συγχρόνω να παραδεχτούμε ότι υπάρχει και μεγάλη πρόοδο. Και αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε, μην το παραβλέπουμε. Σα ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντελβό, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ τον Νίκ Μπαγί, που είχα στο τρένο του και θα μιλήσω γαλλικά. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, με ικανοποίηση σημειώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί την έκθεση της 14ης Μαΐου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβάνοντας μια κοινωνική διάσταση στην οικονομική της πολιτικής, συστάσεις σχετικές με τον περιορισμό του δημοσίου χρέου σε ένα βαθμό θα αντισταθμίζονται από προτάσεις που ενισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικά δικαιώματα και την απόκτηση δεξιοτήτων. Είναι βεβαίως ευπρόσδεκτες οι προτάσεις για την αγορά εργασίας, πολλά όμως ακόμα μένουν να γίνουν για να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και η κοινωνική αδικία είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει συστάσεις για τους μισθούς, την ανισότητα τη μισθολογική, τον προβληματισμό το σχετικό με τους φτωχούς εργαζομένους και τις επισφαλιστές εργασίες. Εάν θέλουμε μια ευρωπαϊκή οικονομία ισχυρή, θέλουμε, πρέπει οπωσδήποτε να βελτιώσουμε τις συνθήκες σχετικές με τους μισθούς. Αυτό άλλωστε έχει προτείνει και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας μεγαλύτερη απασχόληση και ε, ανάκαμψη πιο αποτελεσματική για την οικονομία στο σύνολό τη από ό,τι τώρα βλέπουμε με τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών και των μη μισθολογικών επιβαρύνσεων. Επίσης λοιπόν έτσι μπορούν να περιοριστούν και οι ανισότητες και το κοινωνικό dumping αλλά και να ε, εξασφαλιστεί περισσότερη ευημερία για τα κράτη-μέλη. Ερωτώ εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να ακολουθήσει αυτή την πορεία στα επόμενα χρόνια και θα ήθελα να τοποθετηθώ και στο θέμα των ταμείων συνοχής. Μια φιλόδοξη πολιτική συνοχής μεταξύ κρατών και περιφερειών της Ευρώπης έχει κρίσιμη σημασία. Πρέπει να διατηρήσει την προτεραιότητά της και σε οικονομικούς όρους στον επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυστύχημα το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επαγάγει τμήμα των ε, ευρωπαϊκών κονδυλίων ε, για τη συνοχή στην αιρεσιμότητα του ευρωπαϊκού εξαμήνου πρέπει να είναι αυτόνομη η δυναμική τους και όχι να εξαρτάται από αποφάσεις που λαμβάνονται σε άλλα επίπεδα λήψης αποφάσεων, κάτι το οποίο θα αντέβαινε άλλωστε και στην ε, δυνατότητα για αποδέσμευση και χείρα φέτης των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαχείριση αυτών των κονδύλιων. Ερωτώ λοιπόν γιατί και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να συνδέσει την ερεσιμότητα των, ποσών, των ποσών της συνοχής, των ταμείων της συνοχής με το εξάμεινο και σε ποιο βαθμό αυτό μπορεί να στηρίξει απασχόληση και κοινωνική δικαιοσύνη. Ευχαριστώ κύριος Δομπρόφσκης. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Και καταρχάς θα αναφερθώ στην κοινωνική διάσταση του εξαμήνου. Η Επίτροπος της Ανίδη τοποθετήθηκε εκτεταμένα ήδη όπως είπαμε, ενισχύεται η κοινωνική διάσταση, ενισχύεται, ενσωματώνονται τα ε, στοιχεία τα, κοινωνικού πυλώνα στο εξάμεινο, όπως ανέφερα και νωρίτερα. Ένα τρίτο των συστάσεων και περισσότερο ε, αφορούν ε, την κοινωνική δικαιοσύνη, την αγορά εργασίας και τις δεξιότητες. Επίσης αναφερθήκατε σε μια σειρά αποζητήματα σχετικά με τους μισθούς, την ανισότητα στις συνθήκες εργασίας. Όπως γνωρίζετε με βάση τις αρχές του πυλώνα, του κοινωνικού πυλώνα, έχουμε προχωρήσει σε συγκεκριμένε πρωτοβουλίες και στον τομέα αυτών, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβουλία, αυτό που ονομάζουμε κοινωνική προστασία για τον καθένα, δηλαδή επέκταση της κάλυψης της κοινωνικής πρόνοιας και για τις ατυπικές μορφές ε, της οικονομίας, μορφές εργασίας δηλαδή οι οικονομικές δραστηριότητες, δραστηριότητας που όλο και περισσότερο επεκτείνονται και διαδίδονται. Επίσης έχουμε πρωτοβουλία για το συγκερασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, συνθήκες εργασίας με επικαιροποίηση προηγούμενης ε, ε, δήλωσης επί της οδηγίας και άρα εδώ Μιλούμε όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, αλλά για συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες με στόχο την αντιμετώπιση της απασχόλησης και των κοινωνικών ζητημάτων. Ε, η πολιτική συνοχής και ο συσχετισμός με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όντως, το προτείνουμε για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο με στόχο η ε, να εξεταστεί πώς μπορεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την κοινωνική συμπερίληψη να συνδυαστεί με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και τις συστάσεις αναχώρα. Καθώς έχουμε διαπιστώσει ότι για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις πολύ συχνά χρειάζονται επενδύσεις στα κράτη-μέλη. Βεβαίως, εδώ δεν μπορούμε να πούμε ότι θα είναι απόλυτος και απαρέγκλητος αυτός ο σύνδεσμος υπάρχουν ε, οι προτάσεις ε, στη συνοχή με τους πολύ συγκεκριμένου στόχους. Σε παραδείγματι, στα, στα ταμεία της συνοχής οι στόχοι είναι οι μεταφορές, η ενέργεια, οι υπερβολωτικές υποδομές, οι λοιπές υποδομές και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό κατά πάσα πιθανότητα. Επομένως, ο συσχετισμός με το εξάμεινο θα είναι πιο περιορισμένος. Αφού αναγνωρίζουμε πλήρως ότι η συνοχή έχει ιδίους στόχους να επιτύχει. Και πάνω απ' όλα έχει ρόλο επενδυτικό, ενώ το εξάμεινο καλύπτει διάφορες πτυχές επενδύσεις, διαφορετικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομική πολιτική. Σημειώνω επίσης ότι στο θέμα της συνοχής έχουμε ενισχύσει το μερίδιο του κοινωνικού ταμείου, η SF Plus πλέον έχει γίνει σε μια αιτήσια δέσμη κονδυλίων, αλλά έχουμε συνενώσει και διάφορα ταμεία έτσι ώστε να εξυπηρετήσουμε πιο ικανοποιητικά και αποτελεσματικά ε, τις δράσεις, ιδιαίτερα στην κοινωνική πολιτική, κατά τρόπο ενωμένο, μέσα από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ξεκινήσει, εφόσον εγκρίνουν βέβαια τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι συνομοθέτες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μας πιέζει ο χρόνος και δεν θα έχουμε διερμηνία μετά την προγραμματισμένη λήξη της συνεδρίασης. Ε, γι' αυτό θα ομαδοποιήσουμε τους ομιλητές, αυτό που θα έπρεπε να είχαμε κάνει ήδη από την αρχή. Ε, Έκονη, η δεν βλέπω εδώ τον ομιλητή. Προχωρώ στην ε, Ανθία Μάκεντάιρ, παρακαλώ. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς είναι πολύ καλή είδηση ότι αυξάνονται τα επίπεδα απασχόλησης σε όλη την Ευρώπη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ε, ποσοστό απασχόλησης ρεκόρ και η ανεργία ε, πέφτει συνεχώς, βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο από ό,τι τα τελευταία 40 χρόνια. Ε, οι μισθοί αυξάνονται περισσότερο από τις τιμές, αλλά απομένουν ακόμα πράγματα να γίνουν. Επίσης έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων ε, με... Έχει αυξηθεί το ποσοστό απασχόλησης ανθρώπων με αναπηρίες και Είναι επίσης θετικό ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει αυξηθεί η απασχόληση ατόμων ε, μεταναστών ε, κατά ένα εκατομμύριο. Και όσον αφορά τις συστάσεις αναχώρα για το Ηνωμένο Βασίλειο που αναφέρονται στις δεξιότητες, ε, την τεχνική κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ανθρώπων που βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά γενικά υπάρχει έλλειψη κάποιων δεξιοτήτων ε, και δεν κάνουμε αρκετά ε, στη διδασκαλία των θεμάτων αυτών. Πρόκειται κυρίως για τις θετικές επιστήμες. Τρία λεπτά έχω, διότι μιλώ και για την ΕΚΟΝ και για την ΕΜΠΛ. Εντάξει, τρία λεπτά έχετε τότε, δεν ενημερωθήκαμε. Εντάξει, θα συνεχίσω λοιπόν. Ε, στη χώρα μου έχουμε πάνω από 800.000 καινέ θέσει εργασία. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε οι νέοι να έχουν τι κατάλληλε δεξιότητε ε, για να συμπληρώσουν αυτέ τι θέσει εργασία. Και θα ήθελα να γνωρίζω ε, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το θέμα της επιχειρηματικότητας. Το 85% των νέων ε, θέσεων απασχόλησης προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νεοφυεί επιχειρήσεις. Ε, και τέλος, μιλήσατε για τις ανισότητες. Και θα ήθελα να θίξω το θέμα του χάσματος ε, στις αμοιβέ ανδρών και γυναικών και κατά πόσο το παρακολουθεί αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως και άλλες χώρες, έχουν δεσμευτεί να κλείσουν το χάσμα αυτό που βρίσκεται μέσα στο χαμηλότερο σημείο του από ότι 9,1%. Αλλά θα ήθελα να γνωρίζω τι κάνετε ε, για να λύσετε το πρόβλημα αυτό και πώς παρακολουθείτε την ε, εφαρμογή των μέτρων. Ευχαριστώ. Thank you. So first on, um... Ο κύριος σε ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς όσον αφορά τις ερωτήσεις που σχετίζονται με τις δεξιότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πράγματι έχουμε μία σύσταση για την χώρα σας ε, να αντιμετωπιστεί το θέμα των δεξιοτήτων και να τεθούν ε, στόχοι να εξεταστεί το θέμα των ε, μαθητευομένων και να εξεταστεί το θέμα των δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά τις συστάσεις αυτές για τις δεξιότητες. Ωστόσο, βλέπουμε ακόμα, όπως είπατε, ενώ τα επίπεδα απασχόλησης ε, είναι επίπεδα ρεκόρ όσον αφορά την παραγωγικότητα, φαίνεται ότι δεν εκμεταλλεύονται αρκετά τις δεξιότητες που υπάρχουν και θα πρέπει να εξεταστεί το θέμα της ε, προσληψιμότητας. Στοιχεία του ΟΣΑ δείχνουν ότι το 25% του εργατικού δυναμικού ε, έχουν ε, χαμηλές ή καθόλου δεξιότητες Απομένουν λοιπόν αρκετά να γίνουν ε, όσον αφορά την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη βελτίωση των ευκαιριών ε, και όσον αφορά την ε, τεχνική εκπαίδευση. Αυτή είναι η λογική της σύστασης που έχουμε κάνει. Όσον αφορά την ερώτηση για την επιχειρηματικότητα, σίγουρα αυτό είναι θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, θέματα που έχουν να κάνουν με το επιχειρηματικό περιβάλλον τις δυνατότητες να ξεκινήσει κανείς νέα επιχείρηση, τις δυνατότητες επενδύσεων από πλευρά των επιχειρήσεων, τη δυνατότητά του να δημιουργήσουν νέε θέσει απασχόληση. Αυτά σίγουρα είναι θέματα ευρωπαϊκού εξαμήνου, όπω είναι και το χάσμα στι αμοιβέ ανδρών και γυναικών. Το εξετάζουμε αυτό και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου. Τα κράτη-μέλη με μεγαλύτερη ψαλίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, λαμβάνουν και συστάσεις σχετικά με την, ε, με την μείωση του χάσματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κάρολιν Νατκεκάλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους επιτρόπους που βρίσκονται εδώ σήμερα. Πρόσφατα το Ίδρυμα Μπρίκελ ε, βρήκε ότι όσον αφορά τις συστάσεις αναχώρα, η κατάσταση έχει χειροτερέψει. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένη, η εφαρμογή των μέτρων με ε, μεγάλο έλλειμμα, με υπερβολικό ε, έλλειμμα ε, έχει χειροτερέψει. Τι γίνεται λοιπόν όσον αφορά τις διάφορες χώρες και τους διάφορους τομείς πολιτικής. Ε, και τέλος, έχει βελτιωθεί η εφαρμογή σε κάποια κράτη-μέλη, αλλά γενικά η εφαρμογή των μέτρων ε, συνεχίζει να είναι προβληματική γενικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, πώς θα φροντίσει να γίνουν διαφορετικές μεταρρυθμίσεις, διότι μια σταθερή και ανθεκτική οικονομία είναι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε νέα κρίση. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη που σχετίζεται με αυτήν είναι τα Ευρωπαϊκά Δημοσιονομικά Συμβούλια και το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο πώς μπορούν να συμβάλλουν σε καλύτερο ποσοστό εφαρμογής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ και τον Αντιπρόεδρο που έμεινε μαζί μας για τελειώς γιατί είμαστε εδώ. Πολλά είχα προβλέψει για την κυρία Τάισεν και τον κύριο Μοσκοβισή, αλλά δεν εδώ. Λοιπόν, ακόμα και αν συγκεκριμένα μιλάμε για ένα εξάμεινο αφιερωμένο σε ένα κομμάτι της Ευρώπης, μεγάλη σημασία ποσοτικά και τα λέω στα γαλλικά γιατί θέλω να μιλήσω για την Ευρώπη ακόμα και αν δεν φαίνεται ότι θα το κάνω. Εγώ θα μιλήσω για την Ισπανία, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της Ισπανίας που είναι μια εικονική πραγματικότητα. Για πρώτη φορά ο κύριος Μοσχοβησή υπογράμμισε το πρόβλημα και η κυρία Τίσεν. Δεν κυβερνιέται η Ισπανία σήμερα, είναι διακυβέρνητη. Έχασε την ενή αγορά και όχι μόνο και πολύ περισσότερα από την Ευρώπη σήμερα. Δηλαδή πρόκειται για μια ορολογιακή βόμβα για ολόκληρη την Ευρώπη αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου, το δολάριο, δεν ξέρω τι. Είμαστε στο 18% και οι ανισότητες αυξάνουν και η ανήθικη χρηματοδότηση της κάθε περιφέρειας επίσης αυξάνει. Αδιακυβέρνητη η Ισπανία θα εκραγεί. Συνεπώς, μην κάνετε μόνο την ανάλυση, βάλτε τα όλα, κάντε τα πάντα για να ανακαμφθεί η Ισπανία, αλλιώς θα υπάρχει έκρηξη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Παρακαλώ, απάντηση. Τέσσερα λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Αρχίζω με την υλοποίηση των ειδικών αναχώρας συστάσεων. Αυτό είναι κάτι που Επίσης, θα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την ετήσια προκτική αλλά και την πολιετή. Οι μεταρρυθμίσεις παίρνουν χρόνο, οπότε σε αιτήσια βάση μπορεί να είναι λιγότερο ικανοποιητικά τα πράγματα από ό,τι σε πολιετή. Πάντως όσον αφορά τις εκτιμήσεις μας, οι χώρες μέλη έχουν ή πλήρως υλοποιήσει ή έχουν πετύχει ουσιώδη πρόοδο για το 48 τουλάχιστον των περσινών συστάσεων. Αλλά όντω, η πρόοδος δεν είναι ίδια παντού, ούτε σε όλες τις χώρες, ούτε σε όλους τους κλάδους. Υπάρχουν χώρες με ανισορροπίες, οι μακροοικονομικές ανισορροπίες. Εννοείται ότι η υλοποίηση εκεί δεν έχει προχωρήσει αρκετά όπως σε άλλες. Πάντως σίγουρα πρέπει να υπάρξει περισσότερη πρόοδος. Τώρα συγκεκριμένα τι κάνουμε από αυτού. Ήδη υπογράμμισα κάποια στοιχεία. Κάτι που συχνά λέω είναι ότι εδώ μιλάμε για συστάσεις αναχώρα, έτσι, όχι για διαταγές. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Οπότε κατά πρώτον, αυτό περνάει μέσα από διάλογο και ενστερνισμό ε, της κάθε χώρας των συστάσεων αυτών, ώστε να κάνουν περισσότερο. Προσπαθούμε λοιπόν όσο μπορούμε περισσότερο να είμαστε σε επαφή με τις χώρες για να βελτιωθεί ακριβώς αυτός ο ενστερνισμός. Και δεύτερον, στα πλαίσια του επόμενου πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου, το ανέφερα ήδη, ότι προτείνουμε να ενισχυθεί η σχέση της Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης, Συνοχή και Διευθυντικά Ταμεία, με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Το ρωτήσατε ήδη. Εδώ η πολιτική συνοχή, έτσι κι αλλιώς έχει τους δικούς στόχους, οπότε αυτή η σχέση δεν μπορεί να είναι απόλυτη, αλλά σίγουρα μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες και αυτό ε, το βλέπουμε για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Όσον αφορά το ρόλο τώρα των εθνικών ε, δημοσιονομικών συμβουλίων, αυτά σίγουρα έχουν να παίξουν ένα ρόλο. Και από τη δικιά μας την πλευρά ελέγχουμε και κοιτάμε πώς εφαρμόζουν τις διάφορες διατάξεις οι χώρες μέλη προκειμένου να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν αυτά τα δημοσιονομικά συμβούλια και πώς χρησιμεύουν οι συστάσεις μας και πώς αυτές ενσωματώνονται. Έρχομαι τώρα στη δεύτερη ερώτηση για την Ισπανία. Δεν θα ήμουν τόσο απεσιόδοξος. Η Ισπανία είναι μία από τις ε, μεγάλες χώρες που αναπτύσσονται περισσότερο έχει υλοποιήσει πάρα πολλές μεγάλες μεταρρυθμίσεις την περίοδο μετά την κρίση. Ακριβώ υπογραμμίζουν αυτήν την οικονομική μεγένθηση. Σίγουρα παραμένουν προκλήσεις. Θεωρούμε ότι η Ισπανία εξακολουθεί να έχει μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ε, μεγάλο έλλειμμα, ιδιωτικό και δημόσιο χρέος, χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας. Ε, η ανεργία είπαμε ότι μειώνεται. Πάντως πρέπει να γίνουν περισσότερα, αλλά να σημειώσουμε και την ουσιαστική πρόοδο που έχει πετύχει η Ισπανία μέχρι τώρα. Από την δημοσιονομική άποψη, εγώ έχω ήδη τη γνωμοδότηση για την Ισπανία και φαίνεται ότι συνάδει με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης ε, η Ισπανία και τόσα κάνει και περιορίζει το υπερβολικό έλλειμμα και φέτος. Ευχαριστούμε. Ειρήνα Κάρη. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Επίτροπη, καλώς ορίσατε. Η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016 εισήγαγε τον κοινωνικό πυλώνα το οποίο επενέθηκε και υπόθηκε ότι τώρα πια δεν ε, μας ενδιαφέρει μόνο το κέρδος, μας ενδιαφέρει και η, ε, ε η επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων. Αυτό όμως ε, δεν ταιριάζει πολύ καλά με τις ε, συστάσεις χώρα που βλέπουμε φέτος. Βλέπουμε ότι η Πολωνία, η Μάλτα, η Σλοβενία και άλλες χώρες έχουν αυξήσει το συνταξιδοτικό όριο. Και πολλές από αυτές τις χώρες έχουν πολύ ψηλή ανεργία νέων. Ε, αν αυξήσουμε τώρα την συνταξιδοτική ηλικία θα είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας και γι' αυτό είναι περίεργο από τη μία να έχουμε κοινωνικό πυλώνα που ε, υποτίθεται ότι πρέπει να διασφαλίσει το δικαίωμα στη σύνταξη και να ε, εντάξει τους νέους στην αγορά εργασίας. Ε, από την άλλη όμως βλέπουμε ότι δεν μπορούν να υποφεληθούν από τη σύνταξη αυτή και έτσι υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στον κοινωνικό πυλώνα και τις συστάσεις αναχώρα. Θα λάβετε υπόψη το κοινωνικό πυλώνα στις μελλοντικές συστάσεις αναχώρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς βλέπει τη σχέση ανάμεσα στα δύο θέματα αυτά. Υπάρχει εδώ μια αντίφαση. Πώς θεωρούν λοιπόν ότι θα λειτουργήσει ο κοινωνικός πυλώνας στις συστάσεις αναχώρα. Και τέλος θα ήθελα να ρωτήσω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δείξει μια πιο κοινωνική πτυχή, ε, να μειώσει το σταξιοδοτικό όριο αντί να συνεχίζει να το αυξάνει και να δώσει έτσι τη δυνατότητα στους νέους να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε. Η κυρία και έπρεπε να φύγει, ζητά συγγνώμη. Δεν υπάρχει άλλος από τους πρασίνους. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης λοιπόν τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε Ντομπρόφσκης, ήθελα δύο ερωτήματα να σας απευθύνω. Το πρώτο είναι, καθώς η χώρα μου η Ελλάδα βαδίζει προς την ε, έξοδο, την οριστική από το τρίτο και τελευταίο μνημόνιο, θα ήθελα την δική σας αξιολόγηση για την συμφωνία πακέτο συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων μέτρων ελάφρυσης του χρέους που υιοθέτησε ομόφωνα το Eurogroup πριν μια ακριβώς εβδομάδα, στις 21 Ιουνίου. Πώς την αξιολογείτε εσείς. Και το δεύτερο είναι να σας ρωτήσω γιατί η Ευρωζώνη κατά τη γνώμη σας καθυστερεί και αναβάλει διαρκώς τις αλλαγές που χρειάζεται για να θωρακιστεί απέναντι σε μια μελλοντική κρίση. Ναι, η Ευρωζώνη σήμερα είναι ισχυρότερη από ό,τι ήταν πριν 8 χρόνια, αλλά όχι αρκετά ισχυρή για να αντιμετωπίσει μια νέα κρίση. Και προτάσεις που έχουν κατατεθεί προς αυτή την κατεύθυνση, όπως η ολοκλήρωση τραπεζικής ενοποίησης με την υιοθέτηση του EDIS, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εγγύης Καταθέσεων, ή ένας πιο ισχυρός ESM, ένα ουσιαστικά Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο με ισχυρή δυνατότητα ελέγχου και λογοδοσίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ικανός να απορροφά συστημικά σοκ, διαρκώς παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες. Στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την επόμενη Σύνοδο Κορυφής Ούτε αυτά, ούτε η πρόταση για ένα κοινοτικό, κοινοτικό προϋπολογισμό των κρατών μελών της Ευρωζώνης δεν υπάρχουν στα συμπεράσματα. Γιατί καθυστερεί η Ευρωζώνη να κάνει εκείνες τις αλλαγές ολοκλήρωσης και εμβάθυνσης που είναι απαραίτητες. Η αδράνεια έχει κόστος. Γιατί λοιπόν διαρκώς αναβολές. Thank you. Vice Παρακαλώ, έχετε, να... έχετε το λόγο, την Πρόεδρε, για να απαντήσετε. Καταρχάς, για τις ερωτήσεις που αφορούν το σύνδεσμο και τη διασύνδεση μεταξύ κοινωνικού πυλώνα και ε, συστάσεων αναχώρα. Ήδη έγιναν κάποια σχόλια. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα στο ερώτημα που αφορά τις συντάξεις, την ηλικία της συνταξιοδότησης, δηλαδή ε, σε αντιπαράθεση με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, γιατί υπάρχει πάντα πρέπει να εξασφαλίζουμε εδώ μία ισορροπία. Είναι σαφές ότι καθώς γυράσκει ο πληθυσμός έχουμε ζητήματα βιωσιμότητας μακροπρόθεσμα των συστημάτων συνταξιοδότησης και ε, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Είναι όλο και λιγότεροι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι εργαζόμενοι και σε ηλικία να εργάζονται ε, καλύπτουν τα ταμεία και τις ανάγκες για τις συντάξεις. Μέχρι το 2060 θα είμαστε στο 2 προς 1 Δύο εργαζόμενοι δηλαδή με την εργασία του θα καλύπτουν τι ανάγκε για τη σύνταξη ενό πολίτη. Άρα χρειάζεται μακροπρόθεσμα να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συνταξιδοτικών συστημάτων. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε. Με τη Γενική Αρχή που συνιστά μέσα στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που σημαίνει ταυτόχρονα ότι πρέπει να συνδυαστεί, να συνδεθεί το προσδόκιμο ζωή με το σύστημα το συνταξιδοτικό ε, και να εξασφαλιστεί στο δυνατόν καλύτερη συμμετοχή στην αγορά εργασίας που χρειάζεται για την ε, διατήρηση του κοινωνικού μας μοντέλου. Ε, συγκεκριμένη ερώτηση τώρα που κάνατε για την Ελλάδα. Όντως, έχουμε να κάνουμε με ένα μείζον επίτευγμα. Η Ελλάδα έχει πλέον βγει, βγαίνει από το πρόγραμμα. Εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαιρετίζουμε τις συμφωνίες της 21ης Ιουνίου και τρία είναι τα σημαντικά στοιχεία που θα ήθελα να επισημάνω τώρα για την Ελλάδα. Αφενός μες είναι, πολύ, είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσει την πορεία της ε, στην ε, ε, πορεία για την περίοδο μετά το πρόγραμμα και κυρίως τις διαθροτικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την ευρωπαϊκή οικονομία και κυρίως θα ενισχύσουν την εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή οικονομία για τις αγορές, γιατί τώρα θα στραφεί στις αγορές για χρηματοδότηση η Ελλάδα. Δεύτερον, μέτρα για το χρέος. Επομένως, το πακέτο αυτό για τα μέτρα απομείωσης του χρέους έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η παράταση διάρκειας αποπληρωμής και ε, αναβολή καταβολής του τόκου έχει πολύ μεγάλη σημασία στον περιορισμό του κόστους και εξασφαλίζει ταυτόχρονα πιο σταδιακή, ε, πιο ομαλή, δηλαδή επάνωδο της Ελλάδας στις αγορές. Έχουμε με την συνεχιζόμενη βέβαια του προγράμματος, ε, των όρων μάλλον μετά το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής με το 3% ε, πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι το 2022, ε, μια πιο σταδιακή και μια πιο ανεπτυγμένη, πιο μακροχρόνια δηλαδή, ένα διαμοιρασμό του κόστους χρονικά, μια παράταση δηλαδή του κόστους του χρέους. Ε, υπάρχει ένα ουσιώδες τελευταίο κομμάτι 15 δισεκατομμυρίων ευρώ, αν δεν απατώμε, λέει ο κύριο Ντομπρόφσκη, που έχει να κάνει με ένα μαξιλάρι προστασία για την Ελλάδα, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια σταδιακή και ομαλή επάνωδο στι αγορέ. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Μπορούμε να πούμε πλέον πως η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει στην ανάπτυξη, έχει εξασφαλίσει την οικονομική, τη δημοσιονομική σταθερότητα. Πάνω σε αυτό καλείται τώρα να χτίσει η Ελλάδα και προσδοκία μου είναι πως η ελληνική οικονομία πλέον μπορεί να μας ε, προσφέρει και ευχάριστες εκπλήξεις από εδώ και μπρος. για τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, στο θεματολόγιο και το άνοιγμα του θεματολογίου της ΟΝΕ δεν μπορώ βέβαια να προεξοφλήσω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που είναι εξελίξει αυτές τις μέρες, ωστόσο κάποιες παρατηρήσεις μπορώ να κάνω. Έχουμε κάποια προόδο σε σχέση με την Τραπεζική Ένωση. Από εκεί περιμένουμε συγκεκριμένα βήματα και στοιχεία πιο συγκεκριμένα για, την, ε, για το Ταμείο που έχει ήδη περιγράψει η Επιτροπή και ελπίζουμε ότι το Single Resolution Fund θα το έχουμε λίγο πολύ έτοιμο το Δεκέμβριο. Από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής πρόοδο δεν βλέπουμε ω προ την εγγύηση καταθέσεων Εμεί Θα φέραμε περισσότερο πρόοδο, περισσότερη πρόοδο στον τομέα αυτών. Αλλά ξέρουμε ότι ήταν και ένα θέμα το οποίο προξένησε αρκετέ αντιδράσει από την πρώτη φορά που κατέθεσε την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014. Στα δημοσιονομικά. Και πάλι έχουμε την γαλλο πρωτοβουλία για έναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Εμείς ως Επιτροπή δεν καταθέσαμε πρόταση χωριστή για προϋπολογισμό Ευρωζώνης, αλλά έχουμε χωριστά στοιχεία σημαντικά για προϋπολογισμό Ευρωζώνης μέσα στο προσεχές πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, με την ε, προστασία των επενδύσεων, μάλλον με, το, με τη λειτουργία της σταθεροποίησης και στοιχεία που θεωρούμε ότι είναι συμβατά με τη γαλλογερμανική πρωτοβουλία, αλλά και με πρωτοβουλίε άλλων κρατών μελών. Καθώ στείνουν προς τον ίδιο στόχο, δηλαδή εξασφάλιση ε, μεγαλύτερου περιθωρίου, εργαλείων που θα εξασφαλίσουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο απορρόφησης ε, κλειδονισμών. Και άρα στη συζητήση για τον προπολογισμό περιμένουμε ότι αυτά τα θέματα θα μπουν κυρίως σε όρους πολιτου δημοσιονομικού πλαισίου, γιατί μέσα από αυτό θα προχωρήσουν αυτές οι ιδέες και προτάσεις. Σταματώ εδώ για να δώσει κυρία Τίσεν τι προτάσεις της και απαντήσει τη για το κοινωνικό σκέλος. Ναι, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οπότε κατάλαβα, περιμένετε να σας εξηγήσω τη σχέση ανάμεσα στον κοινωνικό πυλώνα, το κοινωνικό βαθμολόγιο και το εγχείρημα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τι μπορώ να σας πω γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα, στο πυλώνα δεσμευτήκαμε όλοι πέρα αυτού. Έχουμε κάποιες αξίες, κάποιες αρχές, αποτελεί την πηξίδα μας ε, για να ξέρουμε πού θέλουμε να φτάσουμε μαζί. Αν όμως θέλετε να ξέρετε τι κάνετε, πρέπει να μετράτε. Εξού και έχουμε το κοινωνικό βαθμολόγιο, για να μετράμε. Αν δείτε λοιπόν τις ε, συστάσεις αναχώρα και όλα τα έγγραφα τα σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, οι κύριε τάσει του κοινωνικού πυλώνα καλύπτονται. Πρόκειται για πρόσβαση, για ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες, στην κατάρτιση ευκαιρίες για πρόσβαση στην ε, ε, αγορά εργασίας, πρόκειται για συνθήκες εργασίας και πρόκειται και για κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική προστασία για όλους. Αν δείτε τις εκθέσεις αναχώρα και τις συστάσεις, εμπνέονται από τα αποτελέσματα που έχουμε από αυτό το κοινωνικό βαθμολόγιο. Βέβαια δεν θα βρείτε ε, τη λεπτομέρειες για κάθε σημείο, για κάθε χώρα για όλες τις πτυχές. Απλώς εμείς υπογραμμίζουμε που υπάρχουν προβλήματα και χρησιμοποιούμε το βαθμολόγιο αυτό περισσότερο σαν κάποιο screening το οποίο μας επιτρέπει να έχουμε την χοντρική αξιολόγηση αναχώρα μέλος. Τώρα, ξέρουμε ακριβώς χάρη στο βαθμολόγιο που τοποθετείται κάθε χώρα, πόσο μακριά βρίσκεται από τον στόχο προς επίτευξη. Μπορούμε να συγκρίνουμε επίσης την κατάσταση στις διάφορες χώρες μεταξύ τους και τις επιδόσεις τους. Προχωρούν προς τη σωστή κατεύθυνση, κάνουν κάτι λάθος, ε, ποια τα καταφέρνει καλά, ποια τα καταφέρνει λιγότερο καλά και ποια είναι και η συνολική κατάσταση. Είναι ένα καλό εργαλείο που έχουμε στη θέση μας και μας βοηθάει γιατί βλέπουμε αποτελέσματα προκειμένου το ευρωπαϊκό εξάμεινο να γίνει περισσότερο επιτυχές δεδομένου ότι έτσι ελέγχουμε όχι μόνο την οικονομική κατάσταση αλλά και την κοινωνική κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε, Πρόεδρε. Η Λάουρα Αγκαία έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κυρία και κύριε Επίτροπε. Με τις ε, εκτιμήσεις που γίνονται σε σχέση με τις συστάσεις ανακράτος, θα ήθελα να τονίσω ότι η κατάσταση στην ε, Ελλάδα, στην Ιταλία σήμερα δεν φαίνεται να έχει υποφεληθεί από αυτές τις θετικές ε, συνέπειες των μεταρρυθμίσεων, των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων και άρα η αιρεσιμότητα που υποτίθεται ότι θα πρέπει να μπει μέσα στην ε, προσεχή, στον προσεχή δημοσιονομικό σχεδιασμό για την αν, κατανομή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων νομίζω ότι δείχνει μια κάποια δυσκολία ως προς το αποτέλεσμα διότι βλέπουμε από τα στοιχεία τα στατιστικά των τελευταίων ημερών ότι έχουμε 5 εκατομμύρια ανθρώπων στην Ιταλία φτωχών σε επίπεδο απόλυτο, δηλαδή που δεν μπορούν να καλύψουν καν τις, πρωτογεν... τις, πρωταρχικές και κύριες ανάγκες. Ε, δεν καταλαβαίνω όμως γιατί δεν γίνεται μια εκ των προτέρων αξιολόγηση των συνεπειών των μέτρων, γιατί αυτό θα ήταν πάρα πολύ... Παραμένει πολύ ε, επιζήμιο το να μην γίνονται αυτές οι αξιολογήσεις. Βλέπω βεβαίως ότι η Επίτροπος δίνει μεγάλη σημασία στο κοινωνικό περιεχόμενο, αλλά αν δούμε στην ουσία τι σημαίνουν αυτές οι προτάσεις όπως ακούγονται και μάλιστα όπως προκύπτουν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου, η οδηγία για το συγκερασμό του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, αλλά και άλλες οδηγίες μέσα σε μια αρχιτεκτονική που μπορεί να ήταν εξ αρχής ή μάλλον στην αρχή ε, θετική όπως την παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά στη συνέχεια απογυμνώνεται από τα συγκεκριμένα στοιχεία που θα όφιλε να έχει όταν παίρνει από το Συμβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να δω τι είδους προσαρμογές έχετε να προτείνετε. Πρόεδρε επιτρέψτε μου, θα ολοκληρώσω αμέσω. Τι είδους συστάσεις λοιπόν ε, θα κάνετε συγκεκριμένα στο κοινωνικό σκέλος εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μέτρο το οποίο θα πρέπει να δώσει απαντήσεις για το πρόβλημα της φτώχειας, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να εκριζώσουμε τη φτώχεια στην ε, χώρα μας, όπως και παντού. Ταυτόχρονα εγώ νομίζω ότι πάνω απ' όλα πρέπει να φύγει αυτή η αιρεσιμότητα ε, και η, ε, η παγωγή των διαρθρωτικών ταμείων ε, στο εξάμεινο. Ευχαριστώ, Άνεμανς. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Τάισεν. Απευθύνομαι σε εσά. Αναφερθήκατε στα αποτελέσματα χωρών ε, και για το Βέλγιο. Η Επιτροπή μιλάει για ισορροπία του προπολογισμού τώρα αναβάλλεται η απόφαση για το Βέλγιο. Κάθε χρόνο όμως ε, λέτε ότι βελτιώνεται η κατάσταση. Εγώ θα ήθελα να ξέρω να μας το πείτε αυτό συνολικά ε, και τι γίνεται με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Σχεδιασμού που τον Ιούνιο του 2018 είπε ότι το διαρθρωτικό υπόλοιπο αυξάνει, δεν μειώνεται όχι 0,6, ούτε 0,9, αλλά αυξάνεται 4% το 2019 και θα είναι 7% το 2020. Ε, πρόκειται εδώ για το tax shift, όπως ξέρετε. Και ο κύριος Φανροπάου, ο αδερφός δηλαδή του που ξέραμε, λέει ότι φαίνεται να υπάρχει ένας μεγάλος δυναμισμός και ότι δεν θα έπρεπε να σταματήσει με την ε, οικονομική χαλάρωση ο κύριος Δράγκη. Πού βρίσκεται λοιπόν το Βέλγιο τελικά και το χρέος του σε σχέση με την ανακοίνωση αυτή που έκανε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Σχεδιασμού, Οικονομικού Σχεδιασμού του Βελγίου. Ευχαριστώ, Εμίλιαν Πάβελ. Ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ κύριε Τάισεν που επιστρέψατε. Ήθελα μια απάντηση από τον κύριο Γιούνκερ. 14 του μηνός είχα στείλει ένα email και είχατε πει ότι θα ασχοληθείτε με την περίπτωση της Ρουμανίας. Λοιπόν, περιμένω την απάντησή σας στην ερώτηση που έχω στείλει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έρχομαι τώρα στις συστάσεις για τη Ρουμανία. Το 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε 3,6% αύξηση στο ΕΠ. We 7%. Οι διερμηνείς σα ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε στην 24η ημέρα των κινητοποιήσεων και ακόμα δεν έχουμε δει καμία αντίδραση εκ μέρου τη διοίκηση. Αντίθετα, ο Γενικός Γραμματέα κληραίνει ακόμα περισσότερο τη στάση του. Στη σημερινή συνεδρίαση, πολλοί συναδελφοί μα από άλλε καμπίνε έχουν επιταχθεί και είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται. Σε ένδειξη ελληνική, η ελληνική καμπίνα δεν προχωρά σε στάση εργασίας όπως αρχικά προβλεπόταν, ωστόσο η διερμηνία θα διακοπεί ακριβώ τώρα στι 12.30. Ευχαριστούμε και λυπούμαστε πολύ για όλη αυτή την κατάσταση. Wage setting based on objective criteria. Can you define that?